της Λιβύης που δεν του αξίζει η άσχημη αυτή εικόνα την οποία δημιουργούν ορισμένοι ακεραιόφρονες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια αυτή τη Δευτέρα, την 10η Σεπτεμβρίου, μία σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικό μέτρο και μία σύσταση Επιτροπής Γεωργίας περί μη αντίρρησης σε κατεξιοδότηση πράξη δεν εκφράστηκε καμία αντίρρηση στις στάσεις αυτές εντός της 24ωρης προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 87α του κανονισμού. Συνεπώς, οι συστάσεις αυτές θεωρούνται εγκριθήσεις με ισχύ από την 11η Σεπτεμβρίου 2012 και οι αποφάσεις θα δημοσιευθούν σε κείμενα που εγκρίθηκαν τη σημερινή συνόδου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Έλερ, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξ ονόματος όλων των εδώ παρόντων να απευθύνω στην ε, πρεσβεία, στην αντιπροσωπεία καλύτερα των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλους τους εκπροσώπους της χώρας αυτής ε, τα ε, θερμά μας συλληπιτήρια. καταδικάζοντας απερίφραστα αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Απευθύνουμε λοιπόν τα συλληπιτήρια προς των θυμάτων και ιδιαίτερος καλούμε την κυβέρνηση της Λιβύης να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των διπλωματικών αντιπροσωπείων εκεί. Κύριοι συνάδελφοι, η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία της έκθεση κυρίας Παρβάνοβα και της κυρίας Χιμένεθ Μπεσερίλ Μπάριο σχετικά με την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων.